Welcome back. We will now proceed. Καλώς ήρθατε. Και πάλι. Συνεχίζουμε με το σημείο 15 στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Έχουμε επικεντρωθεί πολύ σε αυτό το θέμα για μήνες τώρα. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πυρίνσκι. Παρακαλώ κύριε Πυρίνσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, αυτό το θέμα το έχουμε στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπή μας εδώ και αρκετό καιρό. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας την αξιολόγηση που έχω μέσω των τροπολογιών που υποβλήθηκαν στο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας. Η έκθεσή μου έχει 72 τροπολογίες που προτείνω εγώ όσον αφορά την πρόταση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια υποβλήθησαν 395 τροπολογίες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που μπήκαν στο, σε βάθος σε αυτό το δύσκολο θέμα και να σας παρουσιάσω τις τροπολογίες αυτές. Λοιπόν, 27, 25 συγγνώμη, νές υπάρχουν. Δικές μου, η Άγνες Γιουνκέρης, η Εύελη Ρέγνετ, Μαζί και Σαν Σάιμον έχουν συνυπογράψει. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πιστήσω την προσοχή σας σε τρία ζητήματα αρχής που προέκυψαν διαβάζοντας όλες αυτές τις τροπολογίες και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές για να καταλάβουμε καλά περί τίνος πρόκειται. Το πρώτο στοιχείο έχει να κάνει με την ίδια την φύση λειτουργίας της πλατφόρμας. Τι ακριβώς θα κάνει αυτή η πλατφόρμα. Έχουν ακουστεί ανησυχίες στις διάφορες συζητήσεις μας για το ότι όταν μιλάμε για μέτρα στα πλαίσια της πλατφόρμας υπάρχει αντίληψη ότι η πλατφόρμα θα υπο, θα υπαγορεύει μέτρα. Εξού και ανησυχία πολλών συναδέρφων που αντικατοπτρίζεται και στις τροπολογίες ότι κατά κάποιο τρόπο αφαιρεί προνόμια που έχουν οι χώρες μέλη αυτή τη στιγμή. Το υπογραμμίζω αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι στοιχείο κλειδί για την γενικότερη στάση των χωρών μελών αλλά και των συναδέρφων στην πρόταση αυτή δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας. Όλες οι πλευρές είναι υπέρ. Εκεί που αρχίζουν οι αμφιβολίες είναι όταν ο κόσμος αρχίζει και σκέφτεται μα τι ακριβώς θα κάνει αυτή η πλατφόρμα θα επιβάλλει μέτρα. Εδώ πρέπει να είμαι ξεκάθαρος. Η, η, ιδέα είναι να αποτελεί ένα φόρουμ συζήτησης προκειμένου να ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες ε, πρακτικές, να δίνουμε πληροφορίες υπεύθυνα για αυτήν την ασαφή έννοια της αδήλωτης εργασίας. Και υπάρχουν ποσοτικοί παράμετροι. Τα μέτρα που θα ληφθούν είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να επιβάλλει μέτρα αυτή η πλατφόρμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέρφους, τους σκιώδεις εισηγητές πάνω απ' όλα οι οποίοι συμμετείχαν σε διάφορες συνεδριάσεις που είχαμε τελευταία μάλιστα μόλις χτες. Ο σκοπός ήταν να έχουμε σαφή προσανατολισμό για το περί πρόκειται. Μετά από την παρουσίαση αυτή, μέσα τις επόμενες μέρες, θα προσαρμόσουμε τη διατύπωση έτσι ώστε να παληθεί κάθε αφιβολία που μπορεί να παραμένει για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή αυτή πλατφόρμα δεν επιβάλλει μέτρα. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το θέμα της ε, κανονικότητας. Και άλλες φορές έχω προσπαθήσει να το ξεκαθαρίσω ότι η ευρωπαϊκή αυτή πλατφόρμα πάνω απ' όλα πρέπει να είναι για συνεργασία, πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, για να μην εμφανίζεται αυτή η αδήλωτη εργασία. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια δηλαδή, πρέπει να την αποθαρρύνουμε, να την περιορίζουμε. Συγχρόνως έχουμε μαζική αδήλωτη εργασία που δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε πάρα πολλές χώρες, σχεδόν σε όλες. Οπότε δεν πρέπει να σταθούμε στην αποτροπή, την αδήλωτη και την τιμωρία πρέπει να έχουμε μια επιθετική στάση απέναντι σε αυτήν. Οπότε και εδώ το θέμα αυτό της κανονικότητας, της τακτοποίησης, είναι κάπως ασαφής. Τέλος, αρχόμαστε στο θέμα της ίδιας της λέξης, του νοήματος. Η πλατφόρμα πρέπει να συνεργάζεται ώστε να υπάρχει συμμόρφωση και η αδήλωτη εργασία να μετατρέπεται σε δηλωμένη εργασία. Ήμουν στις γυναίκες τις προάλλες και υποστηρίξαν τον όρο transition, μετάβαση. Πρέπει να το σκεφτούμε τι όρους θα χρησιμοποιήσουμε. Καλό του συναδέλφους και εκείνοι να προτείνουν την καλύτερη δυνατόν διατύπωση, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την έννοια του πώς η αδήλωτη εργασία θα αλλάζει και θα γίνεται δηλωμένη. Το τρίτο θέμα είναι ότι αυτή η ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεν θα είναι ένα φόρουμ για να βγάζει κανείς λόγους. Είναι καλά διαρθρωμένη και σχεδιασμένη έτσι, όπου να λαμβάνει χώρα ουσιαστικός διάλογος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να έχει έναν αρμόδιο που να συνομιλεί και με την κυβέρνηση. Να υπάρχει ένας από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, ένας από τους ευρωπαίους εργοδότες, και θα έπρεπε να δούμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει εδώ. Το θέμα της διαχείρισης τώρα της πλατφόρμας αυτής είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Είδαμε τι γίνεται με άλλες πλατφόρμες, όπου είναι συνδυασμό. Γίνεται διαχείριση με τη συμμετοχή της Κομισιόν από και η αρχή της οικειοποίησης του εστερνισμού γίνεται με όλα τα μέλη της πλατφόρμας. Η βασική ιδέα λοιπόν είναι να έχουμε λειτουργικές κατευθυντήριες γραμμές στην πλατφόρμα ώστε να επιτευχθεί ο τελικός μας στόχος και να δώσουμε προστεθέμενη αξία όσον αφορά την υπευθυνότητα και την υποχρέωση της κάθε χώρας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αδειλώτης εργασίας. Τελειώνω εκφράζοντας την ελπίδα ότι η πλατφόρμα αυτή θα συγκεντρώνει τα συμφέροντα των συνδικάτων, των επιχειρήσεων και των φορολογικών αρχών με την έννοια ότι η πλατφόρμα πρέπει να αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για να τιμωρεί εκείνους οι οποίοι υποφελούνται από την αδήλωτη εργασία, είτε ως δίκτυο, είτε ως επιχειρήσεις που κάνουν ε, στρέβλωση στον ανταγωνισμό με αυτή την τακτική. Πάντως, επίσης, η πλατφόρμα πρέπει να υποστηρίζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων και να μην δέχεται τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας που υφίστανται περισσότερο από αυτούς τους αδήλωτους εργαζομένους. Πρέπει να μπορεί να λειτουργεί καλά η πλατφόρμα και αυτό θα γίνεται εφόσον τονίζουμε ποιες είναι οι καλές πρακτικές. Ευχαριστώ. Περιμένω τα σχόλια των συναδέρφων τώρα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρινσκή. Και τώρα να δώσω το λόγο για δύο λεπτά στους σκιώδεις. Από τα έτη κυρία Ρωμάνα Τόμς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πυρίνσκι για την εργασία που έκανα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έγγραφο αυτό. Και πολλές ήταν και τροπολογίες που έλαβε. Και είμαι σίγουρη ότι πολλή δουλειά ε, έχει ήδη γίνει και πολλοί συμβιβασμοί θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον σε ό,τι αφορά το έγγραφο αυτό. Η ανδρούτη εργασία λοιπόν είναι όντω πολύ σημαντικό πρόβλημα. Σε κάποια κάτι μέλη περισσότερο από ό,τι άλλα, αλλά σε όλα αποτελεί ένα θέμα. Αναγνωρίστηκε ω τέτοιο και από την Λετωνική Προεδρία που το συμπεριέλαβε στις προτεραιότητες της. Και γι' αυτό λοιπόν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε και ένα αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου να αποτραπεί η αδηλωτή εργασία και αυτή η πλατφόρμα αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικά εργαλεία αυτά. Δηλώσουμε ποια είναι τα προβλήματα και στην πολιτική μας ομάδα δώσαμε ιδιαίτερη σημασία σε κάποια από τα θέματα κλειδιά που θα πρέπει να επιληθούν. Αυτό λοιπόν που θα θέλαμε να δούμε είναι το εξή. Ένα πολύ σαφές πλαίσιο για την πλατφόρμα αυτή. Η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο για να επιτυχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι και θα πρέπει να μας επιτρέπει την ανταλλαγή των πρακτικών. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία θεωρούμε που θα πρέπει να επιληθεί ή θα πρέπει να αποτραπεί έστω είναι ότι η πλατφόρμα δεν θα πρέπει να γίνει κάτι που θα έγκυται στην αμμοδιότητα των κρατών μελών. Θα πρέπει να είναι κάτι που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Και είναι βέβαια ότι προ τη σωστή κατεύθυνση κινούμαστε σε σχέση με τι συζητήσει. Και θεωρώ ότι αν ακούσουμε οι μένου δε θα βρούμε ένα καλό συμβασμό προκειμένου το κείμενο να είναι ισορροπημένο στη τελική ανάλυση. Ευχαριστώ. Λίν Μπόιλεν από την QNGL. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. σε συγγήτρια ε, της ΓΚΟΕ δεν μπορεί να έρθει λόγω των ε, προεκλογικών εξωτιών στην Ελλάδα. Πρέπει να επιταχύνουμε την προσπάθεια καταπολέμησης α, ε, της αδίλωτης εργασίας και να αντιμετωπίσουμε αυτό το περίπλοκο φαινόμενο με ευρύ τρόπο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αδίλωτη εργασία έχει πολλές διαστάσεις και πρέπει να τις καταλάβουμε όλες. Γι' αυτό προτείνουμε αλλαγή του ορισμού. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε έναν ορισμό του 1998 που λέει ότι η αδήλωτη εργασία είναι πληρωμένες δραστηριότητες που δεν έχουν όμως ε, δραστηριότητες εργασιακές που δεν έχουν ε, δηλωθεί στις ε, δημόσιες αρχές. Αυτό είναι αφελές. Γιατί μπορεί να έχει δηλωθεί, αλλά μερικώς ε, με πλασματικούς, πλασματικές απολαβές κτλ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις τελευταίες εξελίξεις ε, της αγοράς εργασίας των κρατών μελών. Είναι σημαντικό ούτω ώστε να, δουλε... να προσανατολίσουμε την πλατφόρμα ε, για να μπορεί να ελέγχει το φαινόμενο αυτό. Ε, η ΓΚΟΕ θεωρεί σημαντικό τη σχέση αδίλωτης εργασίας και την ε, πιστοτι... κρίση στα τα τελευταία πέντε χρόνια. Και αναγνωρίζεται τώρα ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην χρηματοπιστωτική κατάσταση στα κράτη-μέλη και τι επιπτώσει που έχει στην άδειλωτη εργασία. Και ένα από τα καθήκοντα τη πλατφόρμα θα, θα πρέπει να είναι εξετάσει αυτή τη σχέση. Τα συμπεράσματα τη πλατφόρμα είναι πολύ σημαντικό ε, για, και μπορεί να επηρεάσει και τα μέτρα λιτότητα. Τώρα, τα μέτρα της ε, πλατφόρμα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ή όχι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σε όλα τα μελη στο βαθμό που δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εσωτερικό κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω την ευαισθησία κάποιων κρατών μελών στο να διατηρήσουν τι αρμοδιότητέ του στο θέμα αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ο αυστηρότερο έλεγχο βλάπτει κάποιον από εμά. Για την νομική βάση ένα σχόλιο θέλω να κάνω, μια και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα τροπολογία των πράσινων ε, με την παραπομπή στο άρθρο 9 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε επίση να υιοθετήσουμε ω άρθρο ε, το αυτό ως ε, νομική βάση. Μια και η κοινωνική ρήτρα της ε, συνθήκης θα πρέπει να είναι ο τόπος όπου εφαρμόζουμε τις κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά και ευχαριστώ τον εισηγητή και ελπίζουμε να συνεργαστούμε καλά στο μέλλον. Τέρι Ράνκε, από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πυρίνσκι για την πολύ εμπεριστατωμένη διαδικασία που ακολούθησε και για τις συναντήσεις με τους σκιώδης συζητητές που είχαμε. Ε, συμφωνώ με την κυρία Τόμς ότι ο αριθμός των τροπολογιών που λάβαμε για αυτή την έκθεση δείχνει τη σημασία που δίνει η Επιτροπή στο θέμα της ατλούτης εργασίας και πολύ ορθά πιστεύω. Δεν υπάρχει μια μία προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικές καταστάσεις και προκλήσεις στα κράτη-μέλη. Όμως η αδίλωτη εργασία εμφανίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή και είναι πρόβλημα και πιστεύουμε ότι η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας θα έχει προσθέμενη αξία για να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα. Μία από τις συζητήσεις που κάναμε αφορούσε την υποχρεωτική συμμετοχή των κρατών μελών και πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα απαραίτητο αυτό. Όχι γιατί θέλουμε να επιβάλλουμε κάτι στα κράτη-μέλη, να είναι τμήμα της πλατφόρμας δηλαδή, αλλά γιατί η λειτουργία της πλατφόρμας εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών και τη θέλησή τους να κάνουν κάτι για αυτό το θέμα στο εσωτερικό τους. Οι πράσινοι θα ήθελαν η πλατφόρμα να περιοριστεί ως προς τα καθηκόντά της, αλλά να έχει σαφέστατη προστιθέμενη αξία και να έχει και εξουσία για αυτά τα θέματα που θα τις αναθέσουμε. Φοβόμαστε ότι αν δεν της δώσουμε την αρμοδιότητα, την εξουσία που χρειάζεται, τότε θα είναι απλώς ένας τόπος συνάντησης και συζήτησης. Και υπάρχουν ούτως ή άλλως ομάδες εμπειρογνωμών που συζητάνε αυτό το θέμα. Θα θέλαμε αυτή η πλατφόρμα να είναι κάτι παραπάνω και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να καταπολεμηθεί αυτό το πρόβλημα της αντιδρούτης εργασίας. Το θέμα της νομικής βάσης ε, αναφέρθηκε από την ΚΟΕ και θέλουμε αυτή η πλατφόρμα στην αρχική της φάση να ξεκινήσει ως πλατφόρμα που τα κράτη-μέλη ε, μιλάνε για τις βέλτιες πρακτικές τους και τις μοιράζονται, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω. Γι' αυτό η αλλαγή της νομικής βάσης θα δείξει ότι αυτό μπορεί να συμβεί και ότι στο μέλλον η πλατφόρμα μπορεί επίσης να παίξει και ένα διαφορετικό ρόλο στην καταπολέμηση αντιλωτής εργασίας. Τελευταίο, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών αναφέρθηκε και είναι σαφής ο προσανατολισμός φύλου. Η κυρία Κούνεβα ήταν η συγγήτρια της Επιτροπής Γυναικών για τη γνωμοδότηση και έκανε πολύ καλές προτάσεις συμπεριλαμβάνοντας και συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το θέμα. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και εμείς όταν μιλάμε για το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Η FTD, Τιτσιάνα Μπέγκη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Πυρίνσκι που είναι εισηγητής τη πρόταση για τον πολύ πλήρη τρόπο με τον οποίο εργάστηκε και εργαστήκαμε. Συμμετείχαμε με μεγάλη επιθυμία έτσι, και όρεξη στις εργασίε, γιατί η καταπολέμηση τη μαύρη και της εργασία είναι πολύ σημαντικό. Το οικονομικό βάρο της πρότασης στον προπολογισμό τη Ένωση είναι αμεληταίο. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν παρόλα αυτά ε, επικαλύψεις με άλλους φορεί ή που έχουν το ίδιο καθήκον. Και μια και μιλάμε για τα λεφτά των φορολογούμενων τη Ευρώπη, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι εξοδεύονται με τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό με τι τροπολογίε μου ήθελα να τονίσω τη σημασία τη πλατφόρμα αυτή, που θα πρέπει να είναι υπεύθυνη απέναντι στην Επιτροπή μα, ούτω ώστε να την ελέγχουμε συνέχεια ότι λειτουργεί σωστά. Ε, Επίση, επιμένω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή λύση και ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μας, όπου η διάσταση και η σοβαρότητα της μαύρης οικονομίας είναι τελείως διαφορετική. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι οι πολιτικές λιτότητας οι οποίες γονάτισαν την Νότια Ευρώπη επιβάρυναν και αύξησαν την μαύρη οικονομία, ειδικά στις χώρες που είναι ενδυμική μάστιγα αυτό. Το να λύσουμε το πρόβλημα της μαύρης οικονομίας, το να βρούμε νέους πόρους για το προπολογισμό των κρατών και να έχουμε περισσότερα δικαιώματα για τους ε, εργαζομένου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ένα πράγμα που θα ήθελα να σα υπενθυμίσω είναι ότι η αντίθετη εργασία δεν ε, γίνεται, αλλά την υφίσταται κανεί. Δεν την κάνει, αλλά την υφίσταται. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την οργάνωση των ακροάσεων που έκανε για να βοηθήσει στην προετοιμασία της έκθεσης. Και κυρίως ευχαριστούμε για τη στήριξη, για τη γενική διάγνωση, στήριξη στην διάγνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να υπάρχει μια ευρωπαϊκή δράση. Ευχαριστώ όλους σας και για τη στήριξή σας στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας. Ξέρουμε ότι τα θέματα του ορισμού θα αποτελέσει αντικείμενο εργασία της ίδια της πλατφόρμας. Οι ορισμοί που προτείναμε αποτελούν μια βάση για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά. Είναι σαφές ότι δεν μιλάμε για παράνομες δραστηριότητες, αλλά, όπως είπε και κάποιος ευρωβουλευτής, υπάρχουν μορφές ψευτοδηλωμένης εργασίας και τέτοιες περιπτώσεις θα εξετάζει η πλατφόρμα. Για το θέμα της ταυτοποίησης. Όντως, είναι ένα ζήτημα που συζητιέται. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά εκτιμούμε ότι το θέμα της νομικής τακτοποίησης είναι απόλυτα θεμητό να εξετάζεται βάσει των πρακτικών στις χώρες μέλη. Κάπου υπάρχουν, όπως στην Ιταλία, ενδιαφέροντα παραδείγματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς, σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις χώρες. Αναρωτιόμαστε κατά πόσο πρέπει να είναι ένας κεντρικός στόχος των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας ή όχι. Αν ναι, μπορεί να εξεταστεί πράγματα στις ανταλλαγές και τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά ίσως και όχι. Να μην πρέπει να είναι κεντρικός στόχος των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας, η οποία για μας, όπως το είπαν και κάποιοι, πρέπει να αποτελεί ένα φόρουμ για να βοηθήσει με πρακτικές λύσεις τους κοινωνικούς εταίρους, στις χώρες μέλη, ή οποιοδήποτε άλλο εταίρο που σχετίζεται με την αδήλωτη εργασία. Να βοηθάει για την ανάλυση και να προσφέρει και συγκεκριμένη συνεργασία. Με επιθεωρήσεις, επιθεωρήσεις όχι μόνο ε, από την επιθεώρηση εργασίας, αλλά και άλλων σωμάτων που να μπορούν να επηρεάσουν την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Έχουμε βέβαια κάποια ερωτήματα για το θέμα της διακυβέρνησης, ναι, όντως, της διαχείρισης δηλαδή της πλατφόρμας. Δεν θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω τα δυνατά σημεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λες και περνώ συνέντευξη για να με προσλάβετε, όχι. Αλλά είμαστε πράγματι σε θέση να συνδέσουμε διαφορετικές ευρωπαϊκές πολιτικές, είτε πρόκειται για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είτε πρόκειται για τη μετανάστευση, τη φορολογία, την εσωτερική αγορά. Όλα αυτά εμείς μπορούμε να τα διαθέσουμε στην πλατφόρμα συνολικά την πραγματογνωμοσύνη μας, δηλαδή και τις εμπειρίες μας για να μπορέσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους και οι διάφοροι Επιπλέον έχουμε και λειτουργικά και οικονομικά μέσα. και τους οργανισμούς που αναφέρονται έτσι καλώς στην έκθεση. Για το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είπε την αρχή ότι θέλει οπωσδήποτε να υπάρχει σύνδεση με τους κοινωνικούς εταίρους. Ίσως όμως να Υπάρχουν και ζητήματα για την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Αυτά για να σας διαφωτίσω λίγο και κατά τα άλλα σας εύχομαι καλή δύναμη για να πετύχετε σε βιβασμό πάνω στην πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πυρίνσκι, τον ε, εισηγητή μας, γιατί θεωρώ ότι με την έκθεσή του κατάφερε να βάλει στοιχεία πολιτικής περισυλλογής για την ανάπτυξη της πλατφόρμας αυτής και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ε, εργαλεία δύο διαστάσεων, αλλά χρειάζεται η συζήτηση να γίνει τριών διαστάσεων. Και θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω για την πολύ σημαντική προσπάθεια που έκανε. Έκανα κάποιες τροπολογίες για να προωθήσω αυτή την ιδέα ίδρυση της πλατφόρμας και να μπορούσουμε να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα ευρωπαϊκό πραγματικά μηχανισμό, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θεωρώ ότι είναι η πιο καλή εφαρμογή της ε, προστιθέμενης αξίας την πλατφόρμα. Η 327, 388, 389 τροπολογίες μου θέλουν να προσθέσουν στην αποστολή της πλατφόρμας αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή τη συμβολή στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για συστάσεις. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένο, προτείνω στα ως προς τα καθήκοντα να υπάρχει κάτι επιπλέον. Η πλατφόρμα να μπορεί να συνδράμει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των ειδήσεων εξαίσεων για την μη δηλωμένη εργασία και την ε, ένταξη των ε, μη δηλωμένων μορφών εργασία ε, στην κανονική και ενόμιμη πλαίσιο. Όλα αυτά να μπουν λοιπόν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, προκειμένου να υπάρχει μια συμβολή και στην ε, ανιούσα και στην κατιούσα φάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στην φάση της δημοσίευσης της έκθεσης της ανάπτυξης, αλλά και στη φάση του διάλογου. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πρακτική και ωφέλιμη πλατφόρμα με τα χαρακτηριστικά αυτά που θα έχει νόημα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν και πάνω από όλα τα κρατημέλη Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάλι τα έχω καταθέσει αυτά στις να εμπλεχθούν και να συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι του ε, δημοσίου τομέα και θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε όλους αυτούς τους τομείς σε βάθος χρόνου. Ευχαριστώ. Γιώργο Μπαλάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε για να προχωρήσει αυτό το θέμα που αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία λόγω της κατάστασης της Ευρώπης και λόγω της εμβέλειας αντίλα της εργασίας. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και εκεί θα επικεντρωθώ. Γιατί ούτε ή πρέπει να φύγω μετά από λίγο. Ισορροπία από τη μία να υπάρχει μια πραγματική πολιτική διαδικασία γύρω από την πλατφόρμα, να υπάρχουν ε, η εταίρια οι απαραίτητη, δηλαδή η κοινωνική εταίρια, αλλά και τα κράτη είναι απαραίτητα να συμμετάσχουν και να μην ε, διαταράξουμε μια πιθανή συνένεση ε, μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να πάμε υπερβολικά μακριά στους στόχους. Γιατί είναι παραγωγικό να είμαστε υπερβολικά, γιατί είναι υπερβολικά ευαίσθητο το θέμα και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και τριβές. Αυτή η μεταρρύθμιση ε, έχει την ανταλλαγή, σαν στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών, την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ότι αφορά την ομιμοποίηση των θέσεων εργασίας. Προσοχή. Σωστά είναι αυτό που λέει η Κομισιόν, ότι μπορεί να είναι ένας από τους στόχους, αλλά όχι ο, ο βασικός στόχος, γιατί ανάλογα με το κράτος για το οποίο μιλάμε, οι πρακτικές είναι διαφορετικές. Και ξέρει ο εισηγητής την γνώμη μου. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με δημοσιονομική ενίσχυση για την νομιμοποίηση αυτών των θέσεων θα ήταν αδιανόητο για ορισμένα κράτη όπως το, δικό μου, ας πούμε. Ε, γι' αυτό μερικέ μερικές τροπολογίες μπορεί να δημιουργούν ρήγη. Γι' αυτό να προχωρήσουμε προσεκτικά. Ρενάτε Βέμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας για τη δουλειά του και υποστηρίζω έντερμα την υποστηρικτή δημιουργία αυτής της πλατφόρμας. Είμαι βέβαια ότι θα ωφελήσει κυρίως τους εργαζόμενους. Όχι μόνο τις αρχές των κρατών μελών να μαζεύουν φόρους, αλλά την προστασία των εργαζομένων στο μέλλον. Κατέθεσα μια σειρά τροπολογιών. Κάποιες ε, στο ίδιο πνεύμα με αυτές και άλλων συναδέλφων, αλλά θα μιλήσω μόνο για λίγα ζητήματα και θα πρέπει να σας πω ότι μιλώ εξ ονόματος, ε, ε μάλλον μιλάω προσωπικά, εκφράζω προσωπική άποψη, όχι την άποψη της ε, Άλτε, τη θέματα των φιλελευθέρων, γιατί απλά πράγματα έχουμε συζητήσει. Κάποια από τα πιο ευαίσθητα θέματα, επιτρέψτε μου να σα δείξω, για την ψευδοαπασχόληση. Θεωρώ ότι αυτή η ψευδοαπασχόληση δεν θα πρέπει να μπει στο πεδίο εφαρμογή που θα καλύπτει αυτή η πλατφόρμα. Δεν είναι αδήλωτη εργασία ουσιαστικά. Είναι μία ανακριβής ε, δήλωση που θα μπορούσε να έχει και μία πτυχή ε, εγκληματική, αλλά είναι στα χέρια των κρατών να το αντιμετωπίσουν αυτό. Ένα άλλο ζήτημα, αντίθετα με από αυτά που έχουμε ακούσει ως τώρα, έχει να κάνει με την υποχρεωτική συμμετοχή των κρατών μελών καταλαβαίνω ασφαλώς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρίσιμο θα έλεγα, να συμμετέχουν όλα τα κρατημέλη στην πλατφόρμα. Διαρωτώ με όμως, με τη νομική βάση που έχουμε στη συνθήκη, μπορούμε να ορίσουμε υποχρεωτική συμμετοχή για τα κράτη-μέλη. Εξέτασα προσεκτικά τη νομική βάση την οποία ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 151-153. Κοιτώντας λοιπόν όλες τις παραγράφους και όλα τα στοιχεία δεν υπάρχει περιθώριο να καταστεί με την οδηγία υποχρεωτική συμμετοχή. Ακόμα και ο ίδιος ο τίτλος μιλάει για ενισχυμένη συνεργασία. Και κοίταξα επίσης το άρθρο 9 το οποίο α, επικαλέστηκαν οι πράσινοι, αλλά αυτό αποτελεί ένα γενικό τμήμα της συνθήκη. Θέλουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να παραμένει στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών και να βρούμε άλλα μέσα να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα αυτή για να μοιραστούν πληροφορίες και ότι όλα θα πρέπει να γίνουν με πάσα σοβαρότητα και τα κράτη-μέλη στη συνέχεια θα κληθούν να αποφασίσουν ε, κατά πόσο θα γίνει αυτό σε περιφερειακό, κεντρικό επίπεδο. Δεν πιστεύω όμως ότι υπάρχει δυνατότητα να ορίσουμε υποχρεωτικό χαρακτήρα συμμετοχής. Ευχαριστώ. Η κυρία Αρένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο για την δουλειά που έκανε Κυρίες, γιατί η πλατφόρμα αυτή είναι πολύ σημαντική για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εργασίας που δεν δηλώνεται σωστά ή δεν δηλώνεται καθόλου. Το θέμα δεν είναι μόνο η ψεύδο ανεξάρτητη είναι η λάθος δήλωση. Είτε πρόκειται για τελώς αδήλωτη, είτε για στραβά δηλωμένη εργασία, πρέπει να καταπολεμηθεί. Και πρέπει να καταπολεμηθεί γιατί αν δεν δηλώνουμε ή δεν δηλώνουμε σωστά κάποιον, δεν τον προστατεύουμε. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και τον αθέμητο ανταγωνισμό. Ο συνάδελφοι από το Άλντε πρέπει να είναι δέστητη σε αυτό το θέμα του ανταγωνισμού. Και το τρίτο, ο λόγος, είναι ότι χάνει χρήματα το κράτος. Τώρα που είμαστε σε λιτότητα, αν μπορούμε να πλουτίσουμε κάπως τα ταμεία του κράτους, θα ήταν πολύ καλό. Κάθε τέτοια πολιτική είναι ευπρόσδεκτη. Συνεπώς, πρέπει όντως να καταπολεμηθεί η αδήλωτη και όχι σωστά δηλωμένη εργασία. Υπάρχουν κάποια θέματα που θα ήθελα να ακουστούν εδώ στο Κοινοβούλιο. Το ένα είναι η συμμετοχή όλων των χωρών μελών. Και ίσως θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο νομικά. Μπορούμε να καταστήσουμε υποχρεωτική αυτή την πλατφόρμα. Πολιτικά νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι η συμμετοχή πρέπει να είναι υποχρεωτική και μάλιστα θα έλεγα πλήρης και ολοκληρωμένη και όχι αλακάρτ όχι ναι, αλλά για μερικά πράγματα μόνο. Όχι. Πρέπει κανείς πραγματικά να θέλει να ανταλλάξει πρακτικές, πληροφορίες από όλες τις χώρες μέλη. Η δεύτερη αρχή, και εδώ συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το θέμα της τακτοποίησης. Δηλαδή, η τακτοποίηση του εργαζόμενου φυσικά είναι κάτι που τίθεται, ξέροντας τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Αλλά η ανησυχία του κύριου Πυρίνσκι είναι κάτι που καταλαβαίνω όταν λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε κατασταλτικά μέτρα. Είναι σημαντικό να έχουμε και μέτρα με κίνητρα, τα οποία να βοηθούν τις χώρες μέλη την άτυπη αδήλωτη εργασία να την κάνουν επίσημη. Δεν πρέπει να προκαταλαμβάνουμε λοιπόν το έργο των χωρών μελών, ναι, και γι' αυτό ίσως να μην αναφέρεται το θέμα της ταυτοποίησης, αλλά να προβλέπουμε τα κίνητρα. Να μην υπάρχει μόνο καταστολή, αλλά να υπάρχουν και κίνητρα. Να βρεθεί το κατάλληλο επιχείρημα που να μας κάνει όλους να συμφωνήσουμε. Τέλος. Πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Η πολιτική συμμετοχή είναι σημαντική βέβαια, αλλά ξέρουμε εμείς οι πολιτικοί ότι χωρίς τις δικήσεις μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Συνεπώς χρειαζόμαστε και αποτελεσματικές διοικήσεις οι οποίες να συνεργάζονται, αλλά χρειαζόμαστε και τους ε, εταίρους μας για να αγωνιστούμε όλοι μαζί κατά της αδήλωτης εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μορβάη. Σας ευχαριστώ, συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι μόνο η αντίλατη εργασία. Η πλατφόρμα αυτή τουλάχιστον δεν θα πρέπει να ασχολείται μόνο με το φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν παρόμοια φαινόμενα. Καταρχάς υπάρχει η αντίλατη εργασία, όπου υπάρχει δηλαδή πραγματικά μια εργασία, υπάρχει εργοδότης, υπάρχει και εργαζόμενος, αλλά ο εργοδότης δεν δηλώνει τον εργαζόμενό του. Και έτσι ο εργαζόμενος δεν έχει κοινωνικά δικαιώματα, δεν λαμβάνει κοινωνικά επιδόματα. Και για παράδειγμα σε περίπτωση παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων τότε μπορεί να στραφεί σε καμία αρχή. Η δεύτερη περίπτωση, το δεύτερο φαινόμενο είναι η ψευδός δηλωμένη εργασία. Οι εργαζόμενοι στην Ουγγαρία, οι εργαζόμενοι αυτοί στην Ουγγαρία έχουν έναν ελάχιστο μισθό που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και στις τροπολογίες ε, αναφέρεται και ένα τρίτο φαινόμενο όπου λόγω φορολογικών ε, πτυχών εξαναγκάζεται ο εργαζόμενος να δηλώσει αυτοαπασχόληση, ενώ στην ουσία δεν είναι αυτοαπασχολούμενος. Και στις τρεις περιπτώσεις λοιπόν αυτός που τελικά α, ε, πλήττεται και είναι εντελώς αυτεθυμένος είναι ο εργαζόμενος ασφαλώς. Ο εργαζόμενος ε, βρίσκεται σε μια καταναγκαστική κατάσταση την οποία δεν έχει επιλέξει και τελικά Στην Ουγγαρία υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, ε, των οποίων μοναδικός στόχος είναι να μεγιστοποιήσουν το, στόχο, το κέρδος τους. Αλλά υπάρχουν και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται στο ότι τα οικονομικά στοιχεία, οι οικονομικές συναλλαγές, οι φορολογικές ρυθμίσεις και γενικά το άχθος είναι τόσο υψηλό που τελικά εξαναγκάζονται να επιλέξουν αυτού του είδους την εργασία. Εμένα μου αρέσει η τροπολογία υπερασμών 91. Εδώ μιλάμε για την επισκόπηση των προλογικών πολιτικών και νομίζω ότι η πλατφόρμα αυτή μεταξύ άλλων θα έπρεπε να έχει και ως καθήκον να καταρτίζει συστάσεις αναχώρα και να εξετάζεται που προκύπτουν οι προβληματικές καταστάσεις σε κάθε κράτος μέλος. Για παράδειγμα, μπορεί ένα κράτος μέλος να κάνει πολλά για τις μικρομεσαίες, αλλά αν η σχετική πολιτική να προκύψει ότι τελικά δεν βοηθούνται επαρκώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή να εξετάσουμε για παράδειγμα το φορολογικό καθεστώ των κοινωνικών επιδομάτων και η πλατφόρμα αυτή θα μπορούσε λοιπόν να πραγματεύεται και τέτοια στοιχεία και ε, το την εισηγητρία κατά πόσο θεωρείται ότι θα μπορούσε η πλατφόρμα να ασχοληθεί και με τέτοια ζητήματα η μη δηλωμένη εργασία και η ψεπτός δηλωμένη εργασία είναι τομεί στου οποίου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανταλλάξουν, να ανταλλάζουν και τι ε, εμπειρίε του και τι γνώσει που έχουν αποκτήσει, τη τεχνογνωσία του, προκειμένου να καταλήξουν σε προτάσει οι οποίε θα προστατεύσουν καλύτερα του εργαζόμενου. Και έτσι να ρυθμιστούν σωστά οι εργασιακές ε, συμβάσει. Σας ευχαριστώ, κύριος ε, Τόμας Μάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και τον εισηγητή ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή βάση από την οποία και προέκυψε ότι η πλατφόρμα αυτή ε, διαθέτει πραγματικά προστιθέμενη αξία, η οποία όμως θα πραγματοποιηθεί αν ε, δεν μείνει σε επίπεδο θεωρητικό, αλλά αν βρούμε τρόπο που πραγματικά μπορεί να βοηθήσουν. Είπαμε στο Κοινοβούλιο ότι Θέλουμε να προωθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, υπάρχει λοιπόν το φαινόμενο της μαύρης εργασίας αλλά και της ψευδός δηλωμένης εργασίας. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμο αναγκάζεται πολλέ φορέ να δεχτεί τέτοια μορφή εργασία, γιατί πολύ απλά δεν έχει επιλογή, αλλά δεν μπορούμε να το δεχτούμε εμεί αυτό. Το είδαμε και στην ε, οδηγία για την απόσπαση, όπου ε, ήταν τόσο έντονα τα μέτρα ελέγχου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίθηκε σε μια διαδικασία διαδικασιών επί παραβίαση. Λοιπόν, δεν μπορείτε να ε, ελέγχετε τόσο πολύ τις εργασιακές συνθήκες και τα κοινωνικά επιδόματα, την κοινωνική προστασία και θέλετε να μεταφραστούν τα έγγραφα στα γερμανικά. Είπαν ε, λοιπόν ότι κάνετε υπερβολικούς ε, ε, ελέγχους. Θα πρέπει όμως αποφάσει το δικαστήριο να γίνεται αυτό. Είναι απαραίτητη η διαφάνεια και από εκεί λοιπόν προς τα αυτή μπορεί να συμβάλλει η πλατφόρμα. Είναι μια πλατφόρμα όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τόσα περιορισμένα ελεκτικά ε, μέτρα, ότι έχουμε τόσους λίγους επιθερητές και να ελπίζουμε ότι θα φτιάξουν από μόνο τους τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενους που έχουν δικαίωμα να έχουν ένα σωστό μισθό. Είναι σημαντικά αυτά. Έκανα λοιπόν μία τροπολογία για να μην μειωθεί σε καμία περίπτωση το επίπεδο ελέγχου. Και η σημαντική σκέψη αυτή, να μην πούμε ότι υπάρχει μια κεντρική, κεντρικοποιημένη αν θέλετε, αρχή, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά τις εμπειρίες αναχώρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μένουν άλλωστε και δικαίως επ' αυτόν οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτά νομίζω ότι πολλές ε, είναι η, συμφων... η συνένεση, μεγάλη συνένεση η οποία έχει προκύψει. Τώρα σε ό,τι αφορά τους όρους θα πρέπει να το κοιτάξουμε, αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση μπορούμε να κάνουμε μια κοινή διαλύωση προς το σωστή κατεύθυνση. Κάποιοι στο Κοινοβούλιο δεν θέλουν να γνωμοδοτήσει, να γνωμοδοτήσουν. Ε, δεν πειράζει, θα γνωμοδοτήσουμε εμείς που έχουμε πάρα πολύ καλή εμπειρία στα τέτοια ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στις εργασίες αυτές και τον ε, εισηγητή. Αυτά που ακούσαμε ήδη είναι πάρα πολύ σημαντικά, εξαιρετικά σημαντικά να δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα και να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό εργαλείο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να τα απαριθμίσω. Επικουρικότητα. Καταρχάς. Πολύ σημαντικό επίσης. Να μην ε, τα βάλουμε όλα στα ίδια καζάνι. Γιατί στα εθνικά κράτη έχουμε σε κάποιο βαθμό πολύ καλά και εύρυθμα λειτουργούσε και λειτουργούνταν και αποτελεσματικά συστήματα. Τα καλά συστήματα λοιπόν που έχουμε σε κάποια κράτη να μην τα αποδυναμώσουμε σε καμία περίπτωση. Δύο-τρία λόγια να πω στις τροπολογίες που έχω καταθέσει. Είναι σαφές, όπως είπα και σε μια προηγούμενη συνεδρίαση, ότι δεν έχουμε ορισμό των κρατών μελών, των, συγγνώμη, της αδελφής εργασίας και αυτό ποικίλει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Γι' αυτό και κατέστησε την τροπολογία υπαρθμών 99 και πιστεύω ότι η πλατφόρμα επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχει να αποτελεί και ένα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων υψηλών βαθμών αξιωματούχων σε θέματα τέτοια. να εκπροσωπούνται οι σχετικοί υπάλληλοι. Αυτό αποτυπώνεται στην τροπολογία υπαριθμό 23. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να διατηρήσουν την αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν τι θα κάνουν σε εθνικό επίπεδο με τα αποτελέσματα της συζήτησης. Και αυτό ε, αποτυπώνται στην 243-244 τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you all for your contribution. Σας ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας. Η οθέτηση στην Επιτροπή Απασχόλησης θα γίνει στις 24 Μαρτίου. Είχαμε μια αρχική ημερομηνία νωρίτερα αλλά έχουμε πολλές ε, συμβαστικές τροπολογίες και χρειαζόμαστε χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Πυρίνσκι <coughs> και ευχαριστώ και τους υπόλοιπους για τη συζήτηση. Και τώρα πάμε στην απαλλαγή, στις απαλλαγές μάλλον. Δώσω το λόγο στην Μαριάν Χάρκιν που είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους. 19 τροπολογίες έλαβα στο σχέδιο γνωμοδοτησής μου. Κατάφερα να δεχτώ πολλές από αυτές και να φτάσω σε συμβιβασμούς. Έχουμε δει τρεις συμβιβασμούς. Ο πρώτος αντικαθιστά την τροπολογία 2, που είναι απλό, απλός. Δεύτερος συμβιβασμός, το συμφωνήσαμε, είναι η 11 και η 13. Και βασικός συμβιβασμός είναι ε, ο συμβασμός που αντικαθιστά τις τροπολογίες 14-18. Θα τα στείλω στους ενδιαφερόμενους όλα αυτά. Ή μάλλον τα έχω στείλει και νομίζω ότι έχουμε συμφωνία. Η μόνη γενική παρατήρηση που θέλω να κάνω για τη γνωμοδότηση είναι ότι έχουμε μικρή μείωση του σφάλματος, του ποσοστού σφάλματος σε όλους τους τομείς. Είναι η χαμηλότερη που είχαμε και το άλλο που πρέπει να τονίσω είναι τα βήματα που έχουν αναλυθεί για να μειώσουμε το ποσοστό σφάλματος ακόμα περισσότερο και κυρίως τα μέτρα που λαμβάνει η Κομισιόν, δηλαδή ε, απλουστευμένες επιλογές κόστους. Αυτή ήταν μία από τις απολογίες που δεν μπορούσα να δεχτώ, που ήταν η 7, όπου είχα γράψει ε, «Καλωσορίζουμε την χρήση των επιλογών αυτών και ο συνάδελφό μου, ο κ. Χολόν, είπε ότι δεν ήταν ε, σύμφωνο. Το ρυθμίσαμε παρόλα αυτά μεταξύ μα. Και τα έργα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν προσθέμενη αξία. Τώρα, στο τέλο μιας περίοδου προγραμματισμού ε, θέλουμε να ξοδέψουμε τα χρήματα, αλλά πρέπει να προσέξουμε, γιατί δεν θέλουμε να Υπάρχει συμβασμό στον αποτελεσματικό έλεγχο, αλλά το βασικότερο είναι α, να έχουν προσ... ειδική προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία τα έργα αυτά και όχι να ξοδεύουμε επειδή απλώ υπάρχουν τα χρήματα. Έπειτα, είμαι ικανοποιημένη με τη δουλειά που έκανε η Κομισιόν και οι αδυναμίες που είχαν ε, εντοπιστεί ε, έχουν αντιμετωπιστεί με κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη-μέλη και υπάρχει πρόοδος σε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να ακούσω την γνωμοδότηση των συναδέλφων. Την γνώμη, συγγνώμη, των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ο σχέδιος ηγητής του ΕΛΚ, ο κ. Χολόν. Πολύ σύντομα, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Είναι μια δουλειά αποτελεσματική προσπαθεί να βρει συμβασμούς η συγγήτρια και να προχωρήσουμε με πολύ αντικειμενικό και προσεκτικό τρόπο. Νομίζω ότι οι συμβασμοί που επετέφθησαν είναι καλοί και δεν θα μας δημιουργήσουν προβλήματα. Και για την τροπολογία 7, το, τη συζητήσαμε ούτως ή άλλως και μπορώ να συμφωνήσω με τη θέση της συζυγήτριας. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα για μας η νομοδότηση και πρέπει να τονίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε για συμβασμούς. Από τους σοσιαλιστές ο κ. Πυρίνσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δουλειά που έκανε η συγγήτρια. Είμαι ευγνώμων που δέχτηκε τις τροπολογίες μου, την 6 και την 19. Συμφωνώ με την προφορική τροπολογία, στην τροπολογία 19 που μας πρότεινε και υποστηρίζω την συμβαστική τροπολογία που συνέταξε η Χάρκιν και που καλεί τις δικές μου τροπολογίες 14 έως 18. Να τη ρωτήσω μόνο. Μήπως μπορεί να εξετάσει αν είναι δυνατόν να έχουμε ένα συμβασμό για τις τροπολογίες 12 και 13 όπου είχα εισάγει μια κάποια διατύπωση, μια κάποια φρασιολογία. Πιστεύω ότι αναφέρονται στα ίδια σημεία. Δηλαδή, ότι η πρόθεση των κρατών μελών όταν απορροφούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να είναι όχι μόνο να τα ελέγχουν αποτελεσματικά, αλλά να πετύχουν και στόχους που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και που είναι σημαντικά πράγματα για τη ζωή κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Το κείμενο που προτείνει η κυρία Χάρκιν λέει το πράγμα αυτό με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει λέει η ανησυχία ότι δεν θα εντοπιστούν οι παραβιάσεις των κανόνων οι κανόνες περί παραβάσεων. Ε, λέμε infringement rules στο αγγλικό κείμενο. Ε, θα έπρεπε να βάλουμε infringement of the rules. Για να είναι σαφές. Παραβίαση των κανόνων. Για τις άλλες τροπολογίες του σχεδίου γνωμοδότησης υποστηρίζω την εισηγήτρια. Τουλάχιστον για τις περισσότερες. 1, 3, 3, 7 και 10. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όλε οι υπόλοιπε υποστηρίζω πλην αυτών που σα προανέφερα, την 1, 3, 7 και 10. Σα ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλε κοιότητε εδώ στη συνεδρίαση. Για σχόλιο, ζητάτε το λόγο. Κυρία Τζεμπάλα, βάλετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία κυρία Χάρκιν και τους σκιώδες και να σας ε, διαβεβαίωσω ότι αναλύσαμε σε βάθος ε, τα θέματα απαλλαγής στην Επιτροπή Κοντ και ήμουν υπεύθυνο και της για τη συγκυρία Τάισεν, την Επιτροπή από την Επιτροπή μας και καταλαβαίνω ε, τη συζήτηση που κάνουν οι συνάδελφοι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό σφάλματο, είναι πιο χαμηλό από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι τα έργα καθίστανται όλο και πιο αποτελεσματικά. Αυτό που εκτίμησα ιδιαίτερω χθε ήταν η συζήτηση για το πώ να διασφαλιστεί ο τελικό αντίκτυπο και ο τελικό προσανατολισμό του έργου. Γιατί αυτό ενδεχομένω να είναι πιο δύσκολο στα κοινωνικά έργα από ό,τι στα υπόλοιπα. Πραγματικά λοιπόν ε, με την Επίτροπο και τους συναδέλφους της εξετάσαμε με λεπτομέρεια το πώς μπορούμε να βρούμε καλούς δείκτες, καλά μέτρα για να προσμετρήσουμε τον τελικό αντίκτυπο, το τελικό αποτέλεσμα. Να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι και οι δύο επιτροπές εργάζονται εξαίρετα για το θέμα αυτό και είμαι πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τα σχόλια από πλευρά τη ε, Επιτροπή ε, Ελέγχου Προπολογισμού. 29 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Απασχόληση, την επόμενη συνεδρίαση δηλαδή. Και έτσι. Αν επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου, λέει η κυρία Χάκη, να κάνω κάποια τελευταία σχόλια. Ναι, θα είναι πάρα πολύ σύντομη. Σας ευχαριστώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και κύριε Πρίνσκι, ναι, ακούω ότι μας λέτε. Έχουμε ανησυχίε. Μπορεί να μπορέσουμε να βρούμε συμβασμό μεταξύ 12 και 13. Ένα άλλο θέμα το οποίο ήθελα να θίξω, θα πρέπει να το έχω θέσει και αυτή εξ αρχή σε ό,τι αφορά την τροπολογία υπερθμών 5. Του συναδέλφου Κάρα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ αλλά νομίζω ότι η αναφορά που γίνεται στην τροπολογία αυτή δεν είναι στακι, δεν είναι ορθή. Το κοινωνικό ταμείο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τι θέσει απασχόληση από ένα κράτο μέλο σε άλλο. Αυτή είναι η ιδέα. Στο, στην αιτιολογική σκέψη υπαριθμών 42 του κανονισμού αναφέρονται μεγάλα έργα. Αλλά όλοι ξέρουμε το ΙΟΣΕΦ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, είναι για επενδύσεις στον κόσμο, στους ανθρώπους, όχι για μεγάλες ε, βιομηχανικές εταιρείε. Καταλαβαίνω το σκοπό της τροπολογίας. Είναι κάτι που απαντάτε στο EGF, απλά δεν είμαι σίγουρη ότι ταιριάζει εδώ και η αναφορά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ορθή. Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σχέση στην προκειμένη περίπτωση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το υποστηρίξει ο πολιτικός, πως υποστηρίζω την ιδέα βεβαίω. Όχι όμως στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν πιστεύω ότι ταιριάζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Μας ικανοποιούν λοιπόν οι απαντήσεις αυτές. Και θα ψηφίσουμε όπως σα είπα στην επόμενη συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 29 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ όλους σας για τις παρεμβάσεις σας.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 των ε, υπηρεσιών. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε λοιπόν το λόγο να δώσουμε και πάλι στην κυρία Χάρκιν. Δεν έχουμε τελειώσει. Ναι, ναι, ναι, μας αγχώνουν και οι πτήσεις επιστροφής. Δεν έχετε ξεμπερδέψει με μένα, αλλά δεν θα μακρηγορήσω. Έτσι κι προχωράμε. Γρήγορα έχω ήδη συζητήσει με τους συναδέλφους, τα έχουμε συμφωνήσει σε ένα μεγάλο βαθμό για τις τροπολογίες. Πρόκειται για τη γνωμοδότηση για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Έχω τρεις τροπολογίες. Και τις τρεις τις δέχομαι, γιατί προσθέτουν θετικά πράγματα στο κείμενο. Και όπως είπα και νωρίτερα, έτσι και εδώ, κοιτάζοντας τα διάφορα έγγραφα, κατάλαβα πόσο καλά δουλεύει το κέντρο. Πιστεύω επίσης ότι το ΣΕΝΤΕΦΟΠ αναγνωρίζεται σαν κέντρο πραγματογνωμοσύνης διεθνώς. Ένα από τα ζητήματα που τίθεται εδώ στη γνωμοδότηση και το έχω συζητήσει και με τους άλλους συζητητές είναι τα επαγγελματικά προσόντα. και σήμερα μάλιστα άκουσα και τη συζήτηση με την κυρία Τάισον. Έχουμε την εντύπωση μερικές φορές ότι χρειάζεται κατάρτιση και αυτό φτάνει. Η τεκμηρίωση το λέει. Πάντως με ικανοποιούν οι τροπολογίες και τις δέχομαι όπως σας είπα όλες γιατί βελτιώνουν το κείμενο. Είσαστε έτοιμοι να περάσετε στο επόμενο. Ή ο κύριος Πυρίνσκι θέλει κάτι να σχολιάσει, παρακαλώ. Μήπως να τις δούμε όλες μαζί τις απαλλαγές, πόσες είναι που μένουν. Να τις κάνουμε όλες μαζί. Συμφωνείτε κύριε Χάρκιν. Παρακαλώ τότε. Καλώς. Ελπίζω να μην πάθω καρδιακή προσβολή. Λοιπόν, για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Βελτίωση εθνικών Διαβίωση και Εργασία. Τέσσερι τροπολογίε είχα εδώ. Και εδώ τι δέχομαι όλε. Γιατί βελτιώνω το κείμενο. Υπάρχει και μια προφορική τροποποίηση. Η τροπολογία αριθμό 2. Δέχομαι. Στη συνέχεια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Τρεις τροπολογίες είχα εδώ. Κάποιες από αυτές ε, όχι πολύ σημαντικές. Η ασυμφωνία με τις Ισπανικές Αρχές για παράδειγμα, ευχαρίστω το δέχομαι. Και η δικιά μου τροπολογία και του κύριου Ρόλαντ. Και εδώ λοιπόν Έχουμε συμφωνήσει τις δέχτηκα όλες. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα επαγγελματική Κατάρτισης τώρα. Δύο τροπολογίες. Η μία είναι δικιά μου και η μία του κύριου Ρόλαντ. Έχουμε μια συμβιβαστική λύση. Τι δέχομαι. Και ο κύριος Ρόλαντ από ξέρω. Αυτά. Αυτές είναι οι άλλες τέσσερις απαλλαγές για τους διάφορους οργανισμούς. Έχουμε δουλέψει καλά, νομίζω ότι συμφωνούν όλοι. Ευχαριστούμε. Mr. Παρακαλώ, κύριε Ρουλά. Ναι, σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ για τις γνωμοδοτήσεις που εξετάζουμε. Όντως, οι συμβαστικές λύσεις είναι θετικές, πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορούμε να τις υποστηρίξουμε χωρίς πρόβλημα. Για τους οργανισμούς, δείχνουμε ότι υπάρχει μείωση του επίπεδου σφάλματος. Έχει γίνει καλή δουλειά επαλήθευσης. Θέλω να προσθέσω όμως και κάποια στοιχεία ακόμα για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Πρέπει να επιμείνουμε. Είναι ένα πολύ καλό κέντρο. Η κατάρτιση είναι ζωτική σημασία σήμερα. Και συμφωνώ με την κυρία Χάρκιν ότι υπάρχει κίνδυνος η μακροχρόνια ανεργία να καταστρέψει τελικά τις δυνατότητες και τα προσόντα που έχουν οι εργαζόμενοι για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Βελτίωσης Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας είναι ένα σημείο αναφορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Πολλές φορές η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στηρίζεται στο έργο του Ίδρυματος αυτού. Και έρευνες που κάνει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας βασίζεται στη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα αυτό για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωση και εργασίας. Είναι οργανισμοί και ιδρύματα δηλαδή πολύ καλά. Και ακόμα και το θέμα της έδρας έχει διαθετηθεί περίπου για όλους τους οργανισμούς. Ο κύριος Πυρίνσκι. κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Χάρκιν και την πρότασή της. Και εμείς δεχόμαστε τις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες αναφέρθηκε. Θεωρούμε ότι όλες είναι καλές. Υπάρχουν κάποια μικρά πραγματάκια που ίσως θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε. Το ένα έχει να κάνει με την έκθεση που αναφέρεται ότι έχει να κάνει με το έργο του Σεντεφόπ. Είναι μια έρευνα που έγινε το 2014 σχετικά με τα προσόντα και θα συζητηθεί στο εκείς μέλλον. Γενικά πάντως είμαστε ευχαριστημένοι. Κύριε Χάρκιν, ευχαριστώ πολύ. Θα συζητήσω μετά με τον συνάδελφο από αυτού. Η τελευταία γνωμοδότηση είναι η απαλλαγή για την εκτέλεση του προπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλους τους οργανισμούς δηλαδή, συνολικά. Επιδόσεις. Εδώ έχω πέντε τροπολογίες, δύο συμβιβαστικές, που πιστεύω ότι τις έχουμε συμφωνήσει, και μία τροπολογία του κ. Πυρίνσκι, την οποία δέχτηκα. Μια στιγμή κάτι ψάχνω ακόμα. Ναι ναι, ένα σχόλιο και θα τελειώσω με αυτό. Μιλάμε για την εφαρμογή της κοινή προσέγγισης όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού κλπ. Είναι σημαντικό να δούμε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος και ότι οι συνέργειες εκεί που επιτυχάνονται, ε, επιτυχάνονται ικανοποιητικά. Κάποιες από τις συμβαστικές τροπολογίες θα δείτε ότι προτείνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί τη δυνατότητα συγχώνευσης οργανισμών. Ξέρω ότι αυτή είναι η άποψη του Κοινοβουλίου, ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό. να υπάρξει συμπληρωματικότητα. Αυτά, κυρία Πρόεδρε. Τίποτα άλλο. Πρόεδρος, ο κύριος Πυρίνσκι. Να ευχαριστήσω και εγώ που δεχτήκατε τις τροπολογίες μου. Και ευχαριστώ για όλη τη δουλειά που έκανε η κυρία Χάρκιν. Ναι, όντω, μια τέτοια δουλειά έχει κινδύνου για την καρδιά μας. Έχετε δίκιο όπως είπατε πριν. Ευχαριστώ και εγώ λέει κυρία Χάρκιν και όλου σας. Τώρα μπορώ να πω ότι έληξε η συνεδρίαση και μπορούμε να επιστρέψουμε στις χώρες μας. Σας ευχαριστώ.